μπορείτε να μπείτε ελεύθερα στο, στο Πακιστάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οποιαδήποτε χώρα, όχι. Ε, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές όπως νομίζει, όπως κρίνει ε, απαραίτητο. Και θα πρέπει οι μετανάστες επίσης να σέβονται τους νόμους της χώρας. Άλλο ο πρόσφυγας ο οποίος προσπαθεί να γλιτώσει τη ζωή του. Αυτούς θα πρέπει να τους δεχτούμε και να τους υποδεχτούμε. Γι' αυτό το λόγο στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να γίνεται η διαλογή, η επιλογή. Ε, μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε το κοινό μας όραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ερώτηση μόνο έχετε δικαίωμα, μία μόνο μπλε κάρτα μπορούμε να δεχτούμε ένα ομιλητή. Οπότε δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλη μπλε κάρτα. Ο λόγος του κύριο Νόιζερ από τους σοσιαλιστές. Κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα με εμένα είναι οι άνθρωποι του οποίου έχουμε ήδη δεχτεί. Έχουμε μια ανθρωπιστική κατάσταση ανάγκης και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην κατάσταση στα νησιά της Ελλάδος. Χρειαζόμαστε αποφασιστική δράση. Το απαιτεί ο ΟΗΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Θεωρώ πως εξευτελιζόμαστε όλοι όταν πρέπει να μα ζητήσει ο ΟΗΕ να δράσουμε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους 12 μήνες. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε ιδιαίτερα την κατάσταση των παιδιών. Ένα τρίτο των όσων φτάνουν στην Ελλάδα είναι παιδιά κάτω των 12 ετών. Και η υγειονομική κατάσταση, όσον αφορά τις αρρώστιες δηλαδή, σε στρατόπεδα τα οποία έχουν ξεχυλήσει, είναι καταστροφική. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως μια διάσκεψη της Κομισιόν της Ελλάδας, της Κροατίας που έχει και την Προεδρία και του ΟΗΕ για να δούμε την κατάσταση στα ε, νησιά και να γίνει ανθρώπινη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάκαρα είναι, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ποιος θα ήθελε να γεμίσει το σπίτι του με κάποιον που δεν κάλεσε. Στη Φιλανδία, στο βορρά, έχουμε την εξή κατάσταση. 35.000 πρόσφυγες μπήκαν, ε, τους λένε πρόσφυγες το 2015 και ως εκ τούτου έχουμε βιασμούς παιδιών και νέων ε, που αυξήθηκαν εκθετικά. Ποιος θα ελέγξει όλα αυτά. Και εμείς έχουμε γυναικόπαιδα στη Φιλανδία. Εγώ πήγα και είδα τα εξωτερικά σύνορα και τους μέτρησα. 500 άνθρωποι, όλοι νεαροί άνδρες. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, λέει, ήταν γυναικόπαιδα. Τα μάτια μου λένε άλλα όμως, δεν λένε ψέματα. Ελπίζω να πούν τα ΜΜΕ την πραγματικότητα. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για ε, κάποιον ο οποίος μπαίνει και κόβει το λαιμό μιας γυναίκης. Ποιος είναι υπεύθυνο. Έχετε μία μπλε κάρτα, την δέχεστε. Ναι, βεβαίως. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Είπατε ότι δεν δεχόμαστε κάποιον στο σπίτι μας που δεν έχουμε καλέσει. Ε, αλλά δεν σας καλέσαμε και σας, αλλά έχετε δικαίωμα να είστε εδώ. Γιατί έχουμε κράτος δικαίου, εκλογικό νόμο και εκλεγήκατε. Και έχουμε ένα σύστημα ασύλου όπου δεν προσκαλούμε κάποιον, αλλά έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να ζητήσουν Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο. Ε, λέτε πραγματικά ότι δεν πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασίες. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Τώρα μιλάμε για εμπόριο ανθρωπίνων όντων. Είναι το ίδιο σαν το εμπόριο ναρκωτικών, μόνο με περισσότερα λεφτά. Και οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Ο κράτος δικαίου δεν σημαίνει ότι ε, δεν μπορούν να διαπράττουν ελεύθερα εγκλήματα. Εκτός αν δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Σας ευχαριστώ. Μπασέσκου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την ελεγμένη μετανάστευση. Αυτό που συμβαίνει ωστόσο μοιάζει περισσότερο με ανεξέλεγκτη μετανάστευση και εμπορία ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύουν από το πρώτο δευτερόλεπτο που φεύγουν από τη χώρα τους. Πρέπει να περάσουν διάφορες χώρες όπου οργανωμένα ε, εγκληματικά δίκτυα τους ε, αναλαμβάνουν για να τους περάσουν από την Μεσόγειο. Είναι υποχρέωσή μας να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση από τη ρίζα της. Χρειάζονται συμφωνίες επανειστοχής, χρειάζονται συμφωνίες όπου οι κυβερνήσεις των χωρών διέλευσης θα εξουδετερώσουν, θα αναλάβουν μάλλον την εξουδετερώση των παράνομων αυτών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και χρειαζόμαστε και ε, ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα σκάφη τα, με τους παράνομους μετανάστες στο λιμάνια προέλευσής τους γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση και θα συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι θα κάνουμε με τα ελληνικά νησιά, με την Κροατία κτλ. Πρέπει να ελέγξουμε τη μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά παρακαλώ να σέβεστε το ένα λεπτό που έχετε ε, χρόνο ε, ομιλίας. Ζήμνιουκ. Σας ευχαριστώ. Ε, συνεχώς μιλάμε εδώ πέρα για μια άλλη τη μεταναστευτική κρίση. Γιατί, Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να δει την πραγματικότητα στα σύνορά της και να αντιδράσει. Συζητάμε γιατί θα κάνουμε τους λεγόμενους πρόσφυγες ε, και μα λέει η βιομηχανία του ασύλου το τι πρέπει να κάνουμε. Πιο μακριά από την πραγματικότητα δεν γίνεται. Δεν είναι δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα. Κλείνουμε τα σύνορα απέναντι σε παράνομους. Άρα και οι βάρκες θα επιστρέφονται ασφαλείς στον τόπο προέλευσης. Θα πρέπει να επιστρέφονται οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα προέλευσης. Αν αρνείται η χώρα να τους δεχτεί πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις αφήνουμε τον κάθε παράνομο χωρίς κανέναν έλεγχο να μπαίνει και ε, απ' την άλλη μιλάτε για φυτογεωνομικά πιστοποιητικά για την εισαγωγή φρούτων όταν φέρνουμε ένα φρούτο από τις διακοπές. Ε, πόσο παράλογο είναι αυτό. Ας στείλουμε επιτέλους το κατάλληλο μήνυμα. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Να εμποδίσουμε τους θανάτους στη Μεσόγειο και το brain drain στις χώρες με ε, να κλείσουμε τα σύνορα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέλη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει και μια πτυχή την οποία δεν έχουμε καλύψει ακόμα. Την οποία αποφεύγουν οι αριστεροί συνάδελφοι και πιο συγκεκριμένα το πώς οι Βόσνοι πολίτες και οι πολίτες των ελληνικών νησιών ζουν το γεγονός ότι εδώ και χρόνια οι μετανάστες ε, περνούν από τα χωριά τους, από τις πόλεις τους ε, ή διαμένουν εκεί και οι ίδιοι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν και από τα σπίτια τους ακόμα. Εγώ είμαι από τη Σερβία και γνωρίζω πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Το 2015 ήταν τόσοι μετανάστες που δεν μπορούσες καν να ζήσεις στο σπίτι σου. Στο νότο της ε, Ευρώπης η κατάσταση χειροτερεύει και θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες ε, πρώτης υποδοχής, δεν είναι πλούσιες χώρες. Ε, επίσης πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες ε, από τις οποίες περνούν οι μετανάστες. Αυτή τη στιγμή είναι φτωχέ χώρε που είναι οι μόνες που φροντίζουν μετανάστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Σιόντροβα από το ΕΛΚ. Κυρίε και κύριοι, η Ευρώπη στα σύνορά της αντιμετωπίζει μια έκτακτη κατάσταση. Η ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων σε ορισμένα hot spot είναι καταστροφική. Εγώ έχω επισκεφθεί τη Μόρια και έχω δει πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Πολλοί από αυτούς μάλιστα δεν έχουν και πού να πάνε, ειδικά αυτοί που προέρχονται από τη Συρία. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τι αιστείε του από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, ε, τη Συρία και άλλα μέρη του κόσμου ε, και ετοιμάζονται να έρθουν στην Ευρώπη. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Οπότε θα συμφωνήσω με τους Κροάτες συναδέλφους. Η κροατική κυβέρνηση και οι Κροάτες συνοριοφύλακες κάνουν ό,τι μπορούν. Πρέπει να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαστε και άνθρωποι και ανθρωπιστές. Και η πιο ευάλωτη ομάδα είναι τα μη συνοδευόμενα, τα συνόδευτα παιδιά. Αυτά πρέπει να προσέξουμε πάνω απ' όλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρέσλερ από το ΕΛΚ. Ο κύριος Ρέσλερ, συγγνώμη. Οι μετανάστες ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως και οι ντόπιοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και είναι φανερό ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση. Οι εικόνες που βλέπουμε από την Ελλάδα είναι πολύ ανησυχητικές. Το ίδιο ισχύει και για τα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2015 υποδεχθήκαμε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, ε, όμως ακόμα και έτσι ε, υπάρχουν καταγγελίες κακομεταχείρισης. Όμως οι αστυνομικοί μας και οι συνοριοφύλακές μας ε, προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της κοινότητας και προστατεύουν τους μετανάστες από κινδύνους. Η Κροατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην υποχωρήσουν εναντί πιέσεων ε, που προσπαθούν, προσπαθούν αυτές οι πιέσεις να αλλάξουν την ε, πολιτική μας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρος, τελειώνει εδώ η συζήτηση. Έχουμε 7 συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο στο πλαίσιο του Catch the Eye. Κλείνει η λίστα. Θα ακούσουμε και τους 7. Λουίς Ντεβέζα από τους Σοσιαλιστές καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ που μας επιτρέπει κύριε Πρόεδρε να πάρουμε όλοι το λόγο, όλοι όσοι τον ζητήσαμε. Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι το ζήτημα αυτό σχετίζεται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα της Ευρώπης. Ε, το συζητάμε επειδή ακριβώ παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα. Όχι μόνο στο σύνορα μεταξύ Κροατία και Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά και αλλού. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στο ύψο των ε, νομικών μας δεσμεύσεων και των αρχών μας. Το είπε και η Κατυπέρη ε, και άλλοι συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι όταν λέει, το, μιλάει το Συμβούλιο για, παράνομες, ε, για παράνομη διάσχυση, ε, Αν όποιο εμφανιστεί στα σύνορα δεν του επιτρέπεται ή δεν του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ασύλου, τι θα κάνει. Αν επιτρέπουμε ταυτόχρονα, ε, αν, δεν επιτρέπουμε επίσης να υποβάλουν αίτηση ασύλου στα προξενία και στις πρεσβείες, πώς περιμένετε ότι θα έρθουν στα εξωτερικά σύνορα να εμφανιστούν και θα υποβάλουν εκεί έτοιμα. Για προσέξτε, για συμπεριφερθείτε λίγο καλύτερα. Παρακαλώ πολύ, ε, τηρήστε την αξιοπρέπεια του, σεβαστείτε την αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Ζόφκο, από το ΕΛΚ, παρακαλώ. reden und die sachen verschieben sich immer weiter nach hinten. das ist eine grobe äh, ε, δεν μας δίνεται σε ποτέ χρόνο να μιλήσουμε και δίνεται συνεχώς το λόγο σε άλλους. Ε, να διευθύνεται σωστά τη συζήτηση. Ένα λεπτό και τέλος. Δεν γίνεται έτσι. Κυρία Ζαύκο, έχετε το λόγο. Ε, είπαμε ότι είναι έντονο το θέμα για μένα γιατί κατάγομαι από τη Βοσνία, πέρασα και τον πόλεμο. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα με αγγίζει. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω τον ε, λόγο τώρα για να μην προκαλέσω περισσότερο τα συναισθήματα. Λοιπόν, Κάποιο κοιμόταν τα τελευταία τρία χρόνια στη Βοσνία, είπε ο Υπουργό των Εσωτερικών. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε τη βοήθεια τη Κροατία και είπε πω η μεταναστευτική κρίση δεν πρέπει να θεωρείται πλέον ανθρωπιστική, αλλά ε, ασφαλεία. Η χώρα χρειάζεται επιγόντως πάνω από 400 επιπλέον ε, συνοριοφύλακες. Από τα 40 εκατομμύρια Ευρωπαϊκή βοήθεια μόνο 7% ε, έχει πάει για τη στήριξη των τοπικών θεσμικών οργάνων τοπικά θεσμικά όργανα τα οποία έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση. Οι μόνοι οι οποίοι ωφελούνται είναι οι διακινητές. Η κροατική αστυνομία συνέλαβε 95 από αυτούς φέτος μόνο. Είναι πανταχού παρόντες, ώστε ο αναπληρωτής διευθυντής της USAID είπε ότι η Αμερική θα κόψει τη βοήθειά της στη Βοσνία εάν δεν σταματήσουν την καταπολέμηση της διακίνησης. Είναι μια ασταθής χώρα. Μην κατηγορείτε τη Βοσνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, να σεβαστείτε το χρόνο. members από την ε, ε, Parliament. Ευχαριστώ. Ε, εμείς οι βουλευτές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα, ειδικά τις βίες αποθήσεις από την Κροατία. Έχουμε τα σύνορα Βοσνίας-Κροατίας που είναι ένα κρίσιμο σημείο, αλλά μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλες μεθορίους, την Γαλλο-Ιταλική ή τα νότια σύνορα της Ισπανίας, όπου έχουμε συχνές αποθήσεις. Πριν από ένα μήνα ε, η Ισπανική ακτοφυλακή επέστρεψε άτομα στο Μαρόκο αφού είχαν φτάσει το Ισπανικό έδαφος, κάτι το οποίο παραβιάζει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και πρέπει να πούμε ότι η συνοριφλακή δεν μπορεί να παραβιάζει τους νόμους και τα ανθρώπινα δικαιώματα επίπλεον. πρέπει να ε, διευκολύνεται το έργο των ΜΚΟ που σώζουν κόσμο όπως το βάσκικο σκάφος το οποίο σε 148 άτομα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γκλάβακ. Γκράβακ από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει. Με την ενίσχυση τη ασφάλεια ε, των πολιτών και μέσω τη πιο αποτελεσματική ε, προστασία των συνόρων, η Κροατία ε, επιθυμεί μια ανθρώπινη συμπεριφορά και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Τα κροατικά σύνορα είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά. Δεν θα σηκώσουμε οδοφράγματα ε, ή εγκαθωτά σύρματα. Ε, όλα όσα κάνουμε στην Κροατία στα σύνορά μας είναι σύμφωνα και συμμορφούνται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα διεθνή στάνταρ. Κροατία καθημερινά έχει άτομα τα οποία θέλουν να περάσουν από το έδαφο τη και, να και να φτάσουν στη Δυτική Ευρώπη. Το μεταναστευτικό πρόβλημα λοιπόν δεν επηρεάζει μόνο μία χώρα αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική μα ιδεολογία δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να διέπεται από ανθρωπιστικέ αξίε. Η μετανάστευση θα πρέπει να είναι ανθρώπινη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, κυρία Αρενά, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ. Το δικαίωμα ασύλου δεν είναι επιλογή, είναι καθήκον. Είναι ένα καθήκον που συνδέεται με τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν το καθεστώς των ε, προσφύγων, βασική αρχή του οποίου είναι η μη ε, επιστροφή και είναι και το άρθρο 2 της συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας και της ισότητας. Η διαχείριση των συνόρων λοιπόν θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συνθήκες και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Ωστόσο, για να περιορίσουμε τις πυρηνιστανευτικές ροές, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σεβάστηκε αυτό το νομικό πλαίσιο και εξωτερήκευσε τη διαχείριση της μετανάστευσης με διμερείς συμφωνίες με χώρες που συχνά δεν πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια ε, για την προστασία των προσφύγων. Όλες οι μαρτυρίες μας λένε πως δεν, είναι, δεν επαρκούν αυτές οι συνθήκες. Εσείς πιστεύετε πως οι δικές μας συμφωνίες αρκούν για το καθεστώς του ε, πρόσφυγες. Πιστεύετε πως ε, το να αναθέτουμε τη διαχείριση μετανάστευση στην Τουρκία, την Βοσνία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ρυθμίζει το θέμα της μετανάστευσης και σέβεται τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, συνάδελφος Κίρτσος του από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθεια που κάνει υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών. Ε, έχουμε φτάσει όμως σε ένα οριακό σημείο, κατά την άποψή μου ε, πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του δουβλίνου για να υπάρξει πιο ανθρώπινη μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών ε, δηλαδή να αλλάξουν οι κανόνες ε, και να, γίνουν, να μοιραστεί το βάρος να μην πέφτει όλο το βάρος στις χώρες πρώτης εισόδου. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι πολιτικά δύσκολο γιατί πολλές χώρες και πολλές κυβερνήσεις είναι σε κατάσταση σοκ μετά την κρίση του 2015-2016 αλλά είναι η μόνη ο μόνος τρόπος να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. επίσης υπάρχει μια πρόταση του έλληνα πρωθυπουργού ε, για τέσσερις χιλιάδες ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν εγκλωβιστεί στην ελλάδα μήπως μπορέσουμε και τους μοιραστούμε στην ευρωπαϊκή ένωση. υπάρχει μια πρώτη ανταπόκριση αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερη. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περέιρα, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί τον εαυτό τη ε, προστάτητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμω ζει μια σημαντική ανθρωπιστική κρίση, όπω αναφέρει και ο ΙΕ. Τα κριτήρια είναι αυστηρότατα και οδηγούν στο να επιλέγουν ορισμένοι και να απορριφθούν άλλοι. Τους κλείνουν όλους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με συνθήκες απάνθρωπες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα οχυρό γύρω της, ε, προστατεύοντας ε, τα, ανθρώπινα, ε, τα εξωτερικά της σύνορα μέσω εγκληματικών συμφωνιών όπως αυτή με την Τουρκία και με άλλες τρίτες χώρες. Επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τη δική της μεταναστευτική πολιτική σε τρίτες χώρες με όπλο την αναπτυξιακή βοήθεια. Μία ακόμα φορά επιμένουμε ότι χρειάζεται να σταματήσει αυτή η παρέμβαση στα εσωτερικά τρίτων χωρών και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο σε θέματα μετανάστευσης. Έτσι τελειώνουμε και το Catch the Eye, οπότε θα δώσω ξανά το λόγο στην Επίτροπο Ντάλι. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Εγώ κρατάω από αυτή τη συζήτηση ότι ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της μη απόθεση όλων των ατόμων είναι προτεραιότητα ανεξαρτήτως του αν είναι εντό ή εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεξαρτήτως αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Συμφωνώ, ότι δεν πρέπει να ασκείται σωματική βία εναντί μεταναστών και προσφύγων και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα τεθούν σε ισχύ τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι, κυρίως τα παιδιά, σε όλα τα στάδια της μεταναστευτικής διαδικασίας. Η αστυνομία και η συνοριοφυλακή θα πρέπει να επιτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι αυτονόητο. Έχουμε αναθεωρήσει την νομοθεσία μας ε, έτσι ώστε να δώσουμε εγγυήσει ε, για την αποφυγή της ε, παραβίασης των θεμελιών δικαιωμάτων. Πρέπει αυτοί οι μηχανισμοί να παίξουν το ρόλο τους. Από τη δική μας πλευρά η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση ε, της δράσης εξωτερικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας και τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μετανάστες ε, από τρίτες χώρες, έτσι ώστε ε, να μην πέφτουν στα χέρια ε, δικτύων διακινητών. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση κ. Ασμάνη, η Κομισιόν θεωρεί ότι οι βασικές προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα συνδέονται εν με την κατά, την εσωτερική κατάσταση των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ θα πρέπει αυτά τα δύο να αντιμετωπιστούν από κοινού. Πολλά από τα θέματα που θίξατε, όπως για παράδειγμα την δευτερογενή μετακίνηση και του συνορικού ελέγχου, ε, τη συνεργασία με τρίτες χώρε και την ανθρωπιστική κατάσταση στα σύνορα, είναι σημαντικά θέματα, κρίσιμα θέματα, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς ε, ενώπιον α, αυτής της ταλαιπωρίας των μεταναστών στα σύνορα. Θα πρέπει από κοινού να διαμορφώσουμε και να διαχειριστούμε την πραγματικότητα της μετανάστευσης. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι μόνιμο πια. Με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας των ατόμων. Και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσετε akkor ε, Ο να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε το θέμα αυτό με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση των μεταναστών, ειδικά των ευπαθών. Γενικότερα, θα ήθελα να επαναλάβω πως η Κροατική Προεδρία θα συνεχίσει να εστιάζει στην εφαρμογή σε σχέση με μια συνολική προσέγγιση του θέματος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά τους πιο αποτελεσματικούς ελέγχους των εξωτερικών συνόρων και να αυξήσουμε την εξωτερική δράση αλλά και τις εσωτερικές πτυχές όσον αφορά αυτά τα οποία ακούγονται για αποθήσεις στα βοσνιακά σύνορα. Όπως όλοι γνωρίζετε, είμαι εδώ πέρα ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν την Κροατία. Θα ήθελα όμως να πω κάτι, γιατί θεωρώ πως ε, η Κροατία αδικείται σε, με αυτούς τους ισχυρισμούς. Υπάρχει μηδενική ανοχή για την βία στην Κροατία. Αυτό το τονίζει η κυβέρνησή μου. και παίρνουμε όλε τι σχετικέ καταγγελίε πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχει καμία άνοχη για καταναγκριστικά μέτρα από την Κροατική αστυνομία κατά οποιοδήποτε και καμία συγκάλυψη οποιοδήποτε αδικήματο που διαπράττουν αστυνομική. Οποιαδήποτε καταγγελία ερευνείται προσεκτικά από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Σα διαβεβαιώ πω η κροατική αστυνομία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των μεταναστών συμμορφούμενοι πλήρω με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Η Κροατία είναι κράτο μέλο της Ένωσης και δρά σύμφωνα με τον κώδικα Σέγγεν και την εθνική νομοθεσία και προστατεύει τα σύνορα και αποτρέπει την παράνομη μετανάστευση. Όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση του κοινού συστήματο ασύλου, παραμένει η προτεραιότητά μας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ευρύτερα και να αναζητήσουμε μια συνολική λύση στι προκλήσει. Έχει γίνει πολλή δουλειά τις προηγούμενες ε, προεδρίες. Και η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να οικοδομούμε στα θεμέλια που έχτισαν. Θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε την ευθύνη με την αλληλεγγύη. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική ατζέντα του Συμβουλίου, η Κροατική Προεδρία ελπίζει ότι το Συμβούλιο αυτό θα αντιμετωπιστεί με το νέο σύμφωνο ε, μετανάστευση και ασύλου και αναμένουμε την παρουσίασή του. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα, είναι μια θετική εξέλιξη το ότι η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα ενέκρινε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για το άσυλο και τα σχετικά ζητήματα όπως ε, οι ε, εγκαταστάσεις ε, υποδοχής. Ετέθη ενισχύει από πρώτης πρώτου. Αναμένουμε την εφαρμογή του. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου έχει μεγάλη σημασία για να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές αλλά και για να εφαρμοστεί η δήλωση με την Τουρκία για τις επανεισδοχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε εδώ η συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Λέγεται καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Νταλή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίγερη αυτή η συζήτηση, γιατί χτε εορτάσαμε την ασφαλή μέρα ίντερνετ σε ολόκληρη την Ευρώπη για 15η φορά μετά από την ε, έναρξη αυτού του εορτασμού το 2014. Θέλουμε τα νέα παιδιά να γίνουν ε, ε, ενήλικες με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, με αυτοπεποίθηση. Το ασφαλές ίντερνετ παραμένει προτεραιότητα γιατί τα παιδιά είναι το 1 τρίτο των χρηστών του ίντερνετ. 8 εκατομμύρια, ε, 800 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν το ίντερνετ Γι' αυτό και είναι μια από τις ε, ε, έξι προτεραιότητες της ε, Κομισιόν να φτιάξει την ψηφιακή Ευρώπη και να επιτρέψει σε όλους και στα παιδιά να ωφεληθούν από την νέα τεχνολογία μέσα σε ασφαλή και δοντολογικά όρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια των ετών με δράσεις που κυμαίνονται από την, ε, το συντονισμό μέχρι την ε, νομοθεσία αυτή καθ' αυτή. τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν και θέλουμε το ίντερνετ να είναι ένα έμπιστο χώρος για τα παιδιά και για όλους τους ε, ανθρώπους. Έχει ξεκινήσει η στρατηγική αυτή το 2012 και έχει συνδυάσει τη συνεργασία κομισιών κατι μέλη η μηχανία της πληροφορικής για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο ίντερνετ για τα παιδιά, συντονισμό αυτό, ρύθμιση και χρηματοδότηση. Η πολιτική μας βασίζεται στην σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου όλα τα κάτι μελη είναι συμβαλόμενα μέρη. Η ασφάλεια, η επικοινωνική ασφάλεια ε, διέπει όλες τις νομοθεσίες σε ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, η νομοθεσία περί σεξουαλικής ε, κατάχρησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, παιδική πορνογραφία και γενικός κανονισμός περί προστασίας των δεδομένων, όπου παρέχονται παντού διατάξεις για να προστατευτούν οι ανήλικοι. Τώρα, στο μέλλον η Κομισιόν θα εργαστεί επί ενός ολοκληρω... μιας ολοκληρωμένης για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και επιγραμμικά. Εκεί θα περιλαμβάνονται δράσεις για να προστατευτούν τα ευάλωτα παιδιά, να προστατευτούν τα δικαιώματά τους online ε, και να ε, προληφθεί και να καταπολεμηθεί η βία. Επίσης θα ενισχύσουμε και θα εξυγχρονίσουμε τους κανόνες που ισχύουν για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση μέσω το... της νομοθεσίας περί ε, ψηφιακών υπηρεσιών θα ε, προσπαθήσουμε να φτιάξουμε σωστή την ισορροπία και να προτείνουμε μέτρα. Επίσης θα καλέσουμε τα κρατημέλη να μεταγράψουν πλήρως ε, την αναθεωρημένη οδηγία περί οπτικοακουστικών μέσων που περιλαμβάνει νέα υποχρέωση για τα κρατημέλη να εξασφαλίζουν ότι οι ε, πλατφόρμες θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα ώστε να προστατεύσουν τους ανήλικους από ε, βλαβερό ε, περιεχόμενο online. Αυτό σημαίνει αναφορά, σήμανση ε, εσφαλμένου περιεχομένου και συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών. Επίσης, η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει ότι τα παιδιά προστατεύονται ακόμα και ε, ε, επίσης για την χρήση των δεδομένων των παιδιών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ούτε για profiling. Το πρόγραμμα δράσης για την ε, ψηφιακή επιμόρφωση θα βοηθήσει τα παιδιά στο να αντιμετωπίσουν την ψηφιακή εποχή. Για να ενθαρρυνθεί αυτό το πρόγραμμα δράσης για την ψηφιακή μόρφωση, θα ενθαρρύνει τα παιδιά και τα σχολεία να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Δηλαδή, ασφαλέστερο ίντερνετ για τις ευρωπαϊκές εκστρατείες, όπου 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι το 2018 και το 2019, όπου καλέσαμε ε, να συμμετέχουν 4,2 ε, εκατομμύρια άνθρωποι 92% από τις 72.000 δραστηριότητες που έγιναν στα σχολεία. Σκοπεύουμε να ενημερώσουμε το πρόγραμμα για να προωθήσουμε την ψηφιακή, το ψηφιακό αλφαβητισμό για τους νέους και τους ενήλικες, ώστε αυτοί να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες που τις χρειάζονται για τη ζωή τους ολόκληρη. Καλύτερο ίντερνετ λοιπόν για τα παιδιά και η Κομισιόν έχει διαβουλευτεί με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να αξιολογήσει τη, το πώς θα είναι ασφαλέστερα τα κέντρα πλατφόρμας ίντερνετ. Η αρχική ανταπόκριση είναι θετική, ε, ώστε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση παρά τους κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση, η κυβερνοπαρενόχληση, ε, ε, ο λόγος μίσους και νέοι τρόποι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Οποιαδήποτε πιθανή ενημέρωση της στρατηγικής θα πρέπει να είναι ε, αρκετά ευέλικτη ώστε να αντέξει και στο μέλλον γιατί το ψηφιακό οικοσύστημα συνεχίζει να εξελίσσεται με τα παιδιά και τους νέους να είναι οι πιο προηγμένοι χρήστε τη τεχνολογία. Τα επόμενα βήματα θα λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα της ε, μελέτης για το πώς οι στρατηγικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη ε, ε, πώς αποδίδουν, τα πορίσματα της διαβούλευσης και επίσης να δούμε πώς θα γίνει η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τις τηλεφωνικές γραμμές, και βεβαίως την εργασία για την νέα στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που ήδη μπορούμε να προβλέψουμε είναι ότι η δουλειά σε αυτό το τομέα θα συνεχίσει να κρατά σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και τη μέτρα ε, χειραφέτησης των νέων και των παιδιών μέσω της, ε, της επίσημης και της ανεπίσημης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος των ομάδων θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Κόπατς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε. Πάνω από 90% των εφήβων στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ από το σπίτι τους. Και μάλιστα είναι η πρώτη ε, γενιά που δεν θυμάται πλέον την αναλογική εποχή. Το ίντερνετ ε, είναι κομμάτι του σύγχρονου κόσμου για τα παιδιά, είτε το θέλουν είτε όχι. Οι νέοι και τα παιδιά αποκτούν τη γνώση τους κυρίως μέσω των τηλεφώνων τους, ε, των ταμπλετών τους ή των λάπτοπ τους. Δεν χρησιμοποιούν σχεδόν πια τυπωμένα βιβλία. Αυτό βέβαια σημαίνει περισσότερη πληροφόρηση και το ίντερνετ ενδεχομένως διευκολύνει και στην εξίσωση των ευκαιριών μεταξύ των παιδιών. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φέρνει και κάποιες απειλές. Δεν είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Ούτε ο, εμείς ως γονείς, αλλά ούτε και τα παιδιά τα ίδια. Συχνά οι γονείς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά μόνοι τους. Ε, και τα παιδιά από την άλλη μεριά αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως το bullying μέσω του ίντερνετ ε, και δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν. Επίσης δημιουργούνται εξαρτήσεις ε, από νέους και παιδιά. Εξάρτηση από τη χρήση του ίντερνετ ή του κινητού τηλεφώνου. Οι προτάσεις για ένα καλύτερο ίντερνετ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ανησυχίες των παιδιών. Ευχαριστώ. Ε, κυρία, ε, κυρία Ντάλη, εκ των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάποτε παρουσίαζα ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα στην τηλεόραση με την ομάδα μου και τότε είχαμε ερευνήσει την ασφάλεια του ίντερνετ για τα παιδιά. Ε, είχαμε βάλαμε ε, μια ψευδή ανακοίνωση ότι ήμασταν 14, μια κορίτσια 14 ετών και τη δημοσιεύσαμε στο ίντερνετ και μετά από ελάχιστες ε, ώρες είχαμε εκατοντάδες άντρες που προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και μάλιστα πολλοί από αυτούς έστειλαν και τα στοιχεία τους προκειμένου να συναντηθούν με το κορίτσι, το δίθεν κορίτσι. Μόλις φτάσαμε εμείς με τις κάμερες ε, άρχισαν να τρέχουν προφανώς. Αλλά βλέπετε πόσο εύκολο είναι ένα παιδί να βρεθεί σε, να πέσει σε μια, μια παγίδα χωρίς να το έχει καταλάβει καν. Τα παιδιά μάλιστα έχουν μια φυσική ε, τάση ε, να αγκαλιάσουν οτιδήποτε είναι στο ίντερνετ. Έτσι εκτίθενται σε πάρα πολλά πράγματα, σε πολλούς κινδύνους, αλλά και σε ψευδείς ειδήσει, σε συγκεκριμένες εμπορικές ή πολιτικές εκστρατείες κλπ. Θα έπρεπε ο ιδιωτικό τομέα, οι κυβερνήσει και οι γονεί να προσπαθήσουν από κοινού να προστατεύσουν τα παιδιά και θα πρέπει ε, το ίντερνετ να γίνει ασφαλές για τα παιδιά. Με τον ίδιο τρόπο που θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή στο σχολείο, στο δρόμο. Έτσι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή και στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Renew Europe, η κυρία Τόμ έχει το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε εκδήλωσε ενδιαφέρον να μιλήσω ε, στο θέμα αυτό γιατί ήμουν εισηγήτρια σχετική έκθεση. Οπότε διάβασα τα σχετικά και απογοητεύτηκα όταν είδα ότι η τελευταία φορά απασχόλησε την Κομισιόν το θέμα το 2011 και έκτοτε το ξεχάσαμε. Πριν από 10 χρόνια ήμασταν κατά του κατακαιρματισμού της αγοράς. Πριν από 2 χρόνια όμως εγκρίναμε την λεγόμενη ηθική ανάπτυξη των παιδών που θα ορίσουν τα κράτη-μέλη. Το 2019 η Κομισιόν ανακοίνωσε την σύσταση μιας ομάδας ειδικών. Οπότε μόλις 8 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει το πρώτο βήμα. Έκτοτε η ομάδα συνεδρίασε 3. Αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί καμιά λύση. Γιατί υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και πρέπει να δράσουμε αναλόγω. Δέκα χρόνια για μια πολιτική απόφαση σημαίνει μια γενιά που πέρασε. Δεύτερον, δεν μπορούμε να λύσουμε συστημικά προβλήματα με έργα. Ναι, έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρθηκαν ε, κατά πολέμηση σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης, ξενοφοβίας κτλ. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να υπάρξει ψηφιακή εκπαίδευση των παιδιών ε, σε κάθε σχολείο. Υποχρεωτικά, με καλούς δασκάλους, σωστό, σωστή ύλη και αξιολόγηση. Τι έχουμε στην πράξη, κάποια κράτη-μέλη όπου 60% των σχολείων δεν είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Ε, τι λέμε τότε. Θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να επενδύσουμε και να δώσουμε λεφτά όχι στις συνεδριάσεις εδώ πέρα, αλλά στα σχολεία. Αλλιώ σε άλλα δέκα χρόνια τα ίδια θα λέμε. Σας ευχαριστώ. Από το ID τον λόγο έχει ο κύριος Φέστ. Ναι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε όταν εμφανίζεται κάποιο σφάλμα στον ορίζοντα, αμέσως υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι η αυξημένη χρήση του ίντερνετ οδηγεί σε μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης, τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να γράφουν και γίνονται ακόμα και πιο παχύσαρκα. Και δεν μιλάμε καν για το περιεχόμενο του ίντερνετ. Ε, είτε μιλάμε για grooming, ε, ε, είτε πορνογραφία και ψευδείς ειδήσει. Δεν θα πρέπει να προωθούμε τη χρήση του ίντερνετ ε, από το παιδιό, γιατί ακόμα και τα αθώα ηλίθια παιχνίδια τα εμποδίζουν να συγκεντρώνονται και να κάνουν άλλα σημαντικότερα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να βοηθάει τον κλάδο να παγιδεύει τους καταναλωτές όλο και νεότερους όπως προστατεύουμε τα παιδιά από το αλκοόλ και την πορνογραφία, πρέπει να τα προστατεύουμε και από αυτή την αποβλάκωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κόλαγε από τους πράσινους. Έχει τον λόγο. Το ασφαλές ίντερνετ για τα παιδιά είναι κρίσιμο. Τα παιδιά θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλή και θα πρέπει να διατρήσουν την περιέργεια τους, να ανακαλύψουν πράγματα. Όμως έχοντας κοιτάξει το, τη σελίδα στο ίντερνετ της μέρας για το πιο ασφαλές ίντερνετ ε, διαπίστωσα ότι οι συζητήσεις εστιάζουν στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί υλικό που έχει σχέση με τις σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ε, εμείς ε, αναλύουμε και πρέπει να αναλύσουμε τα θετικά και τα αρνητικά αυτών των τεχνολογιών και γι' αυτό το λόγο είναι λίγο πρόωρο να σκεφτούμε ε, την, το, να, να πιστέψουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα ότι ε, θα, ε, μάλλον θα προτιμούσα να εστιάσουμε στην εκπαίδευση. Οι μελλοντικέ πρωτοβουλίες της Κομισιόν θα πρέπει πράγματι να εστιάσουν στην ανάπτυξη των, ε, της, των τεχνικών ικανοτήτων των παιδιών και τη επιμόρφωσης τους έτσι ώστε να μπορούν να προστατευτούν. Ευχαριστώ. Μόλις τη Γκουε η κυρία Πελετιέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. 75% των παιδιών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που ανοίγει παράθυρα σε άλλους κόσμους όμως είναι και ένα πεδίο κινδύνων. Έχετε δίκιο, Επιτροπή, που λέτε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας που αντιμετωπίζουν κινδύνους. Και χαίρομαι ε, για τον, την καταπολέμηση της, ε, του, εγκλήματος, του, ε, του του, και άλλων φαινομένων που πλήττουν τα παιδιά στο ίντερνετ. Όμως, στην ανακοίνωσή σας λυπάστε που οι νέοι καταναλώνουν στο ίντερνετ. Ε, έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία του ίντερνετ που σπρώχνουν τους νέους στην κατανάλωση. Στην ανακοίνωσή σας, την οποία έχω εδώ στα χέρια μου τέλος, ε, ζητάτε ένα ψηφιακό κόσμο για όλους. Εσείς πρέπει να βελτιώσετε την κατάσταση και την ζωή των ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, που έχουν αναπηρίες κλπ. Για αυτούς δεν λέτε τίποτα. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να μιλήσετε για ένα ψηφιακό κόσμο που δεν θα ξέρει κανέναν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπυράκη τώρα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Εξ του ΕΛΚΑ. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε είμαι σίγουρη ότι ξέρετε ότι η μισή από τους νέους έντεκα έως δεκαέξι ετών στην ευρώπη έχουν εκτεθεί σε έναν από τους βασικούς κινδύνους του διαδικτύου cyberbullying sexting online grooming ή fake news. ως πρέσβυρα για το ασφαλές διαδίκτυο για όλους κάνω στην ελλάδα εκδηλώσεις ενημέρωσης των μαθητών και τους ζητάω να μας δείξουν πώς προστατεύονται όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα είναι θεαματικά τα παιδιά μας είναι υποψιασμένα. όμως χρειάζονται βοήθεια και η βοήθεια πρέπει να έρθει από εμά και πρέπει να έρθει με την επιστράτευση της τεχνολογίας. όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εφαρμογές του διαδικτύου είτε αυτές είναι παιχνίδια είτε αυτές είναι social media έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να εντοπίσουν προβληματικό υλικό στο διαδίκτυο που απευθύνεται για παιδιά να εντοπίσουν παρενοχλήσεις και να τις διακόψουν νομίζω πως εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση στη χρηματοδότησή τους. ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενημέρωση των δασκάλων των γονέων και τελικά των παιδιών. πρέπει να προστατεύσουμε τους ψηφιακούς πολίτες του αύριο. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το επιγραμμικό περιβάλλον είναι σημαντικό χώρο ζωή. Μπορεί να είναι και ένα χώρο συμμετοχή και χειραφέτηση, όπω δείχνει για παράδειγμα ε, τα Fridays for the Future. Ε, ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο επιγραμμικός κόσμος είναι ασφαλής για τα παιδιά. Ορισμένα φαινόμενα είναι, ε, μπαίνουν αυξανόμενα, όπως οι διάφορε διακρίσει, η διάδοση πορνογραφικού υλικού, ε, έκθεση σε πορνογραφία, κυβερνο παρενόχληση. Πρόκειται για σοβαρέ βλάβε στου ανηλίκου. Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα ε, μέσα πρόληψη πέρα από την εκπαίδευση, πριν από την ε, γνωστική χρήση του ίντερνετ. Ε, μπορούμε να ενισχύσουμε τα μέσα ε, εντοπισμού και αφαίρεση συγκεκριμένου υλικού από το διαδίκτυο. Στην προηγούμενη θητή είχαμε υποβάλει εδώ στο Στρασβούργο μάλιστα μία πρόταση νομοθεστήματος που εγκρίθηκε στην Ιταλία ακριβώς για την κυβερνοπαρενόχληση και είναι πολύ σημαντική και επί της ουσίας. Πρέπει λοιπόν οι νομοθέτες, η βιομηχανία και η κοινωνία των πολιτών να ασχοληθούμε και να εστιάσουμε ειδικά στην ε, ανάθεση ευθυνών σε όλους και στην ε, ε, αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ως νομοθέτες σε ένα περιβάλλον επιγραμμικό που να είναι ασφαλές. Πρέπει να είναι άμεση μας προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Ρέσλερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των παιδιών από την επιγραμμική κατάχρηση. Το ίντερνετ είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που δίνει τεράστιες ευκαιρίες, όμως υπάρχουν εκεί και κάποιοι κίνδυνοι. Μόνο με τις, σωστέ ασφαλιστικέ ε, σωστές μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και να τους προστατεύσουμε από το λόγο μίσος, ε, την παραπλανητική διαφήμιση και την κυβερνοπαρενόχληση. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν οι τεχνολογικές εταιρείες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί. Ωστόσο, θα πρέπει εμείς να έχουμε τον ε, ρόλο της ασφαλιστικής δικλίδας μαζί με τους γονείς που αυτοί, σε αυτούς τρέχονται τα παιδιά όταν έχουν προβλήματα στο ε, διαδίκτυο. Εμείς θα πρέπει να εργαστούμε για ένα ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον που τα παιδιά με ασφάλεια αυξάνουν τις γνώσεις τους, την επικοινωνία τους και τις συνδέσεις τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ακίου Σαλίμπα είναι ο επόμενος ομιλητής εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών. Ενώ το ίντερνετ προσφέρει πολλές ευκαιρίες, δημιουργεί και κάποιους κινδύνους, ειδικά στις πιο ευαίσθητους, ευάλωτους χρήστες και κυρίως τα παιδιά. Στον διαδικτυακό κόσμο, τα παιδιά εκτίθενται συχνά σε βλαβερό και παράνομο περιβάλλον. Και υφίστανται ε, σεξουαλική ε, κακοποίηση, ε, πορνογραφικό υλικό, βλέπουν πορνογραφικό υλικό κλπ. Στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται με πολλούς τρόπους τα παιδιά, μαθαίνουν, παίζουν κλπ. Και θα πρέπει ε, να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν βέβαια κίνδυνοι όπως υπάρχουν κίνδυνοι, είναι φυσικό να υπάρχουν κίνδυνοι όπως υπάρχουν κίνδυνοι και στον εξωτερικό κόσμο. Όμως θα πρέπει να τους δώσουμε τα κατάλληλα προσόντα και ταυτόχρονα να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτούν. η ηθική μας ευθύνη, ηθικό μας καθήκον να τους προσφέρουμε ένα πιο ασφαλές ίντερνετ. Η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένες αποτελεσματικές ε, εγγύησεις ε, για αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιμπουρόπουλος, παρακαλώ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου χθε και ως ψυχίατρος αντισυχώ, κυρία Επίτροπε. Μόνο στην Ελλάδα ένα στα πέντε παιδιά έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης 60% έχει μπει σε ακατάλληλο περιεχόμενο, εκτεθειμένα σε ρητορική μίσου, σε ψυχολογικέ επιθέσει, σε εκβιασμού και σε οικονομικέ απάτε. Τα μισά παιδιά δηλώνουν ότι αυτό τα έβλεψε ψυχολογικά και τα όθησε σε κοινωνική απομόνωση. Πολλοί γονεί αφήνουν τα παιδιά με το κινητό στο χέρι. Η εξάρτηση των παιδιών τα κάνει ευάλωτα, επιθετικά και τα απομονώνει. Το διαδίκτυο δεν είναι παιχνίδι. Χρειαζόμαστε σύγχρονη παιδεία που οχυρώνει τα παιδιά από αυτού του κινδύνου. Πρέπει να εξαναγκάσουμε τους παρόχους και τι εταιρείε λογισμικού για να εξασφαλίσουμε δωρεάν ή τουλάχιστον πολύ φθηνό λογισμικό προστασία των παιδιών. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενημερωμένων Ευρωπαίων γονέων να μπορούν να καταφύγουν σε μια εύχρηστη διαθέσιμη ευρωπαϊκή εργολιοθήκη. Χρειάζεται να γνωστοποιήσουμε τον χρόνο και τον τρόπο τη υγιού χρήση του διαδικτύου Πρόκειται για δίκοπο μαχαίρι που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε από τι αρνητικέ και επιδικίνδυνε συνέπειέ του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κλείνουμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μιλητών και περνάμε στη διαδικασία του Catch με έξι συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα τους ικανοποιήσουμε και τους έξι. Καταρχήν, ο κ. Νεγκρέσκου, του μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να χτίσουμε ένα ασφαλές ίντερνετ για τα παιδιά μας. Σε συνεργασία με, με αυτούς που δίνουν περιβάλλον, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους παρόχους κλπ. Μια πρόσφατη μελέτη στην Ρουμανία έδειξε ότι ένα στα τρία παιδιά σε ηλικίε 9-16 υφίσταται κυβερνομπούλινγκ και είναι ένα φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται. Σχεδόν τα μισά από τα παρενοχλημένα παιδιά δεν έκαναν τίποτα. Δεν αντέδρασαν. Γι' αυτό το λόγο μερικές φορές οι και μάλιστα μερικές φορές οι ενήλικες δημοσιεύουν ιδιωτικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία των παιδιών τους στο ίντερνετ, χωρίς να καταλαβαίνουν τι κακό μπορούν να κάνουν. Θα πρέπει να στηρίξει η Κομισιόν την ψηφιακή εκπαίδευση και αυτή όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες και για τους γονείς και για τους δασκάλους. Είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτή από την Κομισιόν και είμαι πεπισμένο ότι το ίντερνετ θα γίνει ασφαλές αν το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το πολύ. Κύριε Λουκα... από το ΕΛΚ. Οι έρευνες σε πολλές χώρες δείχνουν ότι ε, όλο και πιο μικρά τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το σταματήσουμε. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι λένε ότι παιδιά δεν κοινωνικοποιούνται επαρκώς εξαιτίας ε, της υπερβολικής ε, απασχόλησής τους με το ίντερνετ. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τουλάχιστον να είναι ασφαλή στο ίντερνετ και ότι το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση να είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία τους. Έχουν, υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τους νέους στο ίντερνετ, αλλά υπάρχει και η πορνογραφία, η ρητορική μίσους, το μόμπινγκ, η παιδοφιλία, η, ε, η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση κλπ. Θα πρέπει επίσης να γίνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού ε, για τους κινδύνους οι οποίοι, ε, τους οποίους ενέχει η χρήση του ίντερνετ και Ελπίζω η Κομισιόν να μπορέσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να κάνει το ίντερνετ ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χάιζερ από τους σοσιαλιστές. Κύριος Χάιζερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην ε, Σλοβακία λέμε ότι το ίντερνετ είναι σαν τη φωτιά είναι καλός υπηρέτης αλλά κακός αφέντης. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να ξεφορτωνόμαστε τα παιδιά με το να τους δίνουμε μία ταμπλέτα ή ένα τηλέφωνο. Όχι, πρέπει να γίνει το ίντερνετ όμως ασφαλές για τα παιδιά μας ε, και πρέπει βεβαίως ε, να προστατεύουμε τα δεδομένα των παιδιών, να μην πέφτουν στα δίχτυα παιδεραστών ή εταιριών, γιατί τα παιδιά βλέπουν πολλές διαφημίσεις ε, στο διαδίκτυο ή μέχρι και σεξουαλικές απαφές. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί με τους γονείς και τα σχολεία για να υπάρξει ένα πρόγραμμα εκπαίδευση στο ίντερνετ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως ε, υπάρχει και δουλειά των ε, γονιών και των σχολείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να παλέψουμε στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν χρειάζεται νομίζω να περιγράψω όλους τους κινδύνους, τις πρακτικές, ε, ε, όλους τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Συμφωνώ πως η εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας είναι ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο για να βελτιώσουμε την προστασία των παιδιών και εμείς ως ευρωβουλευτές πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόζεται σωστά στα κράτη-μέλη. Όμως το αποτελεσματικότερο εργαλείο είναι η πρόληψη και αυτό σημαίνει να διδάσκουμε τα παιδιά να φέρονται σωστά. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους, ε, τους γονείς που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τα παιδιά και εδώ πέρα θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να σας πω το εξή. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα που αναπτύσσουν τα πανεπιστήμια μας ε, στην Τσεχία π.χ. Το πανεπιστήμιο